Αγαπητοί συνάδελφοι, ε, ε, ας ε, αρχίσουμε τη συνεδρίασή μας για σήμερα το απόγευμα. Το πρώτο σημείο είναι το σημείο 12. Έκθεση του Καρλ Σλάιτερ, ρυθμιστικές πτυχές των ανοηλικών. Καρλ, θέλεις το λόγο ή να περάσουμε κατευθείαν στην ψηφοφορία. Όχι, θέλεις το λόγο. Ε, ξέρετε, ε, είναι νέο αυτό το θέμα, διότι οι πολιτικές ομάδες δυσκολεύτηκαν να συντονίσουν τη θέση τους. Ε, δυσκολευτήκαμε πολύ στις διαπραγματεύσεις, γιατί ενώ είχαμε συμφωνήσει στην αρχή, μετά αλλάξαμε, άλλαξαν κάποιοι γνώμοι, συνεχώς αλλάζαμε τη στάση τη γραμμή που θα ακολουθούσαμε όλοι από πλευρά όλων των πολιτικών ομάδων δυσκολευτήκαμε γιατί είναι καινούριο σχετικά το θέμα αυτό και δεν έχουμε πάγιες θέσεις αν θέλετε, τις διαμορφώνουμε κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Ελπίζω να γίνουν δεκτές οι συμβαστικές λύσεις που βρήκαμε οι φιλελεύθεροι δεν δέχονται πλέον την ενοποιημένη τροπολογία υπαριθμών 19. Αλλά αυτό είναι ατυχές, διότι αν δεν πούμε τίποτα για το ότι η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν καλύπτει επαρκώς ε, τις ανάγκες που υπάρχουν ε, για την νομοθετική ρύθμιση, ε, τότε τροποποιούμε την ίδια την αρχή της έκθεσης. Οπότε ε, ζητώ από τους συναδέλφους σε προσωπικό επίπεδο να επανεξετάσουν αυτή την ενοποιημένη τροπολογία γιατί στην αρχή υπήρχε ευρεία υποστήριξη και μετά σταδιακά απέσυραν όλη την αποστήριξή τους και είναι πάρα πολύ δύσκολη μια τελευταία έκκληση που απευθύνω στους συναδέλφους αλλιώς να αρχίσουμε την ψηφοφορία. Ε, γιατί έχουμε τις και τις ε, συμβαστικές τροπολογίες ε, και ουσιαστικά θα διεξαχθεί πολύ γρήγορα η ψηφοφορία. Αλλά για λόγους συνέπειας, καλό είναι να επανεξετάσουν οι συνάδελφοι τη θέση τους. Θέλουμε να είμαστε λίγο πιο ουδέτεροι στις δηλώσεις περί νανοτεχνολογίας και θέλουμε να υπάρχει μια ευρεία βάση, ευρεία αποδοχή. Νομίζω ε, με αυτόν τον τρόπο θα περάσουμε το σωστό μήνυμα. Τι θέλει το Κοινοβούλιο χωρίς όμως ε, ε, να, ε, να πούμε ξεκάθαρα ακριβώς τι θέλει το Κοινοβούλιο δηλαδή. Ωραία, ας περάσουμε στην ψηφοφορία. Έχετε την, τον κατάλογο των ψηφοφορίων, έχετε τις κάρτες σας. Συμβαστική 1 και 2 μαζί τις ψηφίζουμε. Ποιοι είναι υπέρ παρακαλώ κατά αποχές ε, εγκρίνεται. Συμβαστική 3, 4, 5, 6, 7 ομαδών υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. Ενοποιημένη 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Συμβαστική 9 υπέρ κατά, αποχές, εγκρίθηκε. Συμβαστική 10, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε. Συμβαστική 11, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε. Συμβαστική 12 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίθηκε Ενοποιημένη τροπολογία 13. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εξακρίβωση παρακαλώ ηλεκτρονική. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 19 υπέρ, 10 κατά, εγκρίθηκε λοιπόν. Συμβαστική 14 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίθηκε. Ενοποιημένη 15 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίθηκε. Συμβαστική 16 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται ενοποιημένη 17 ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ενοποιημένη 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ενοποιημένη 19 υπέρ κατά αποχές ε, εξακρίβως ηλεκτρονική Έρχεται η ψηφοφορία για την 19, υπενθυμίζω. Ψηφίστε παρακαλώ. Είμαι πολύ υπομονητικός. Λίγα δευτερόλεπτα ακόμη. Πέρας ψηφοφορία, ζητώ συγγνώμη. 17 υπέρ, 13 κατά, εγκρίθηκε. Ενοποιημένη 20 υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω με την ίδια πλειοψηφία εγκρίθηκε. Ε, συμβαστική 21 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ενοποιημένη 22 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ενοποιημένη 23 υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ενωποιημένη 24 υπέρ, κατά, Εξακρίβωση, παρακαλώ, επαλήθευση ηλεκτρονική. Ψηφίστε, παρακαλώ. Για την 24, υπενθυμίζω. Ηλεκτρονική ψηφοφορία έχει ανοίξει ήδη, έχει αρχίσει η ψηφοφορία και τώρα Τελειώνει. 17 υπέρ 13 κατά. Εγκρίθηκε όντω. Συμβαστική 25. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ενοποιημένη 26. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ενοποιημένη 27. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ενωπημένη 28. Αυτή έχει αποσυρθεί. Πάμε στην 29. Υπέρ. Κατά. Επαλήθευση παρακαλώ. Την 29. Επαληθεύουμε για την 29. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας η ίδια πλειοψηφία 17, 17 ψήφι προς 13. Εγκρίθηκε. Συμβαστική 30 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 31 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 32 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 33 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 34. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ενοποιημένη 35. Υπέρ. Κατά. Νομίζω με την ίδια πλειοψηφία θα εγκριθεί, αλλά επαλήθευση παρακαλώ. Για την 35 ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Νομίζω είναι η ίδια πλειοψηφία πέρας, 17 ψήφι προς 13. Ε, εγκρίθηκε. Λοιπόν, θα ε, σας πω ποιες ε, τροπολογίες καταπίπτουν επειδή εγκρίθηκαν σε αυτές οι συμβαστικές και ενοποιημένες τροπολογίες. Employment, Επιτροπή Απασχόληση 7, στη σελίδα 5 στο δικό μου κατάλογο. Ελπίζω να βρήκατε όλη την τροπολογία αυτή. Ποιοι είναι υπέρ παρακαλώ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε. Ε, τροπολογία 90, Βέστλουντ, υπέρ κατά ένα λεπτάκι να, κάνω μια να κάνουμε την επαλήθευση ηλεκτρονικά την 90 έτσι Βέστλουντ. Νομίζω θα είναι 17 προς 14 τώρα. Ε. Διαδικαστικό. Λυπάμαι πάρα πολύ. Θα ήθελα να ψηφίσω υπέρ, αλλά έχασα την κάρτα μου. Κοίταξα κάτω. Ε, λοιπόν, ζήτησα από τους τεχνικούς να μου δώσουν μια άλλη κάρτα. Λυπάμαι, δεν ξέρω τι έγινε η κάρτα μου. Θέλω πάρα πολύ να λάβω μέρος σε αυτή την ψηφοφορία, αλλά δεν ξέρω τι να κάνω. Λυπάμαι πάρα πολύ. Ε, το, τα γερμανικά μου είναι πολύ φτωχά, αλλά καταλαβαίνω ότι χάσατε την κάρτα σας. Ε, τι μπορούμε να κάνουμε. Ίσως είναι προσωπικό σας πρόβλημα. Μπορείτε να έχετε μία επιπρόσθετη κάρτα ή, κάτι, ή κάτι τέλο πάντων. Υπάρχουν μερικές τεχνικές ε, δυνατότητες. Λοιπόν, ε, κατά τα άλλα είναι αδύνατο. Αδύνατο. Είναι παρούσα, είναι παρούσα. Λυπάμαι πάρα πολύ. Υπάρχουν ορισμένοι κανόνες και λυπάμαι πάρα πολύ. Λοιπόν, λοιπόν, σας παρακαλώ, αν θέλετε να πάρετε το λόγο για διαδικαστικό, σηκώστε το χέρι σας. Λοιπόν, υπάρχει μια διαδικασία και έχουμε αποφασίσει πάνω σε αυτό το θέμα σχετικά με την ηλεκτρονική ψηφοφορία δεν είναι δυνατόν να σηκώσετε το χέρι σας και να αντικατασταθεί με αυτόν τον τρόπο ε, η παρουσία σας, η ψήφο σας τη στιγμή που υπάρχει ηλεκτρονική ψηφοφορία. Λοιπόν, λοιπόν τροπολογία 19. 90. 17 προς 14 ε, λοιπόν για την τροπολογία 90 βέσλοντ. 78 του ο κ. Σλάιντερ, ποιοι είναι υπέρ κατά Αποχές εγκρίνεται. 79 Καρσλάιτερ υπέρ. Κατά. Αποχές. 17 προς 14 δεν είναι πάλι. Άντε, επαλήθευση, ηλεκτρονική επαλήθευση. Oh, there is one additional member present κατέφθασε κι άλλος ένας βουλευτής, θα αλλάξουν τα νούμερα. 17 προς 15 θα έχουμε τώρα. Λοιπόν, πέρας ψηφοφορίας. Α, 16 προς 15. Ναι, αλλά εγκρίθηκε. 68 Φερέιρα, υπέρ. Κατά. Ξανά λοιπόν, ξανά, ξανά. Ε, ε ηλεκτρονικά ψηφίστε. Την 68 Φερέιρα παρακαλώ. Άρχεται η ψηφοφορία. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά την 68. Πέρας. 16 προς 17. καλω ήρθατε κυρία Κουτιέρες Κορτίνες λοιπόν. Ε, 80, 80 σλάιτερ υπέρ, κατά, ηλεκτρονική επαλήθευση. Everybody had voted. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. 17 προς 16. Εγκρίνεται. 81 Slater υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονική επαλήθευση. Άρχεται. Η ψηφοφορία. Πέρας. 16 προς 17. Απερίφθη. Ο αντιπρόεδρος Μπλόκλαντ είναι ε, ε, ε, VIP βλέπω. Ε, τρία της Επιτροπής Απασχόλησης υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η δέκα της Επιτροπής Απασχόλησης υπέρ. Κατά. Ποχές. Εγκρίνεται. Η 82 σλάιτερ υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονική επαλήθευση. Την 82 ελέγχουμε έτσι. Πέρας. Ψηφίσατε όλοι, ε, ελπίζω. 19 προς 16. Εγκρίθηκε. 13 της Επιτροπής Απασχόλησης. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Με διαφορετική πλειοψηφία ηλεκτρονική επαλήφθηση. παρακαλώ. Για τη 13, έτσι, της Επιτροπής Απασχόλησης. Ψηφίσει ηλεκτρονικά. Πέρας. 22 προς 13 εγκρίθηκε. 14 της Επιτροπής Απασχόλησης υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονική επαλήθευση. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. 18 προς 17. Εγκρίθηκε. 88 σύνοτ υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονική επαλήθευση. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρασε 21 ψήφι προς 13. Εγκρίθηκε. 106 Φερέιρα. Ποιοι είναι Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονική απαλήθευση. Ψηφίστε. Ηλεκτρονικά. Πέρας. 17 προς 16 εγκρίνεται. 93 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονική επαλήθευση. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας. 21 ε, ψήφι προς 13 εγκρίθηκε. 94 τώρα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ε, σχεδόν ταυτόσημες 96-97 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνονται. 95 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Ναι, 98 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Εντάξει, θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά την 98. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας. 9 προς 24, όντως ε, απορρίπτεται. Εκατόν ένα Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Ποχές. Εγκρίνεται. 102 ρις υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται.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 Και τώρα κάνω ένα τεράστιο άλμα και πάω στην επόμενη σελίδα, 9 δηλαδή. Δύο ταυτόσημες έχουμε, 19 και 20. 19 και 20 διότι στους φακέλους σας λέει ότι καταπίπτει, καταπίπτει λόγω της έγκρισης της ενοποιημένης 28 αλλά δεν εγκρίθηκε ενοποιημένη 28 οπότε πρέπει να τις ψηφίσουμε οπότε υπέρ για 19 και 20. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Απορρίπτονται και οι δύο. 21 λίτερ υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 30 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. 31 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονική επαλήθευση. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας, 18 προς 17. Εγκρίθηκε. 34, λίτερ υπέρ. Κατά. ίδια κατάσταση, ηλεκτρονική επαλήθευση λοιπόν για να είμαστε σίγουροι. Πέρας. 18 προς 17 εγκρίθηκε. 35 υπέρ. Κάτα. Αποχές. Εγκρίνεται. 43 σλίτερ υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Επαλήθευση 43. Πέρας. 30 προς 5. Εγκρίθηκε. 44 υπέρ. Κατά. Αποχές. Επαλήθευση. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρασε. 17 προς 18 περίφθη Ο κύριος Μπλόκλαν το αποφάσισε αυτό. 45 υπέρ. Κατά. Αποχές. Επαλήθευση. Ψηφίστε. Πέρας. 17 προς 17 ισοψηφία απορρίπτεται. 46 υπέρ. Κατά. Αποχές. Επαλήθευση. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας. 17 προς 18.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 Πέρας. 21 προς 14. Εγκρίθηκε. Ευχαριστούμε, Κάσλιτερ. Συγχαρητήρια κιόλας. Τώρα πάμε στο 14. Επιτροπολογία, καταχώρηση, αξιολόγηση, αδειοδότηση και περιορισμή των χημικών προϊόντων. Το ρίτσι δηλαδή. Ο Σα... κύριος Σακώνη θα πάρει το λόγο. Και μετά πρέπει να ψηφίσουμε την ε, προφορική ερώτηση και το σχέδιο ψηφίσματος. Κύριε Σακώνη. My dear ε, ε, σας παρακαλώ, προχωρούμε στο επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης και σας παρακαλώ πολύ επιτρέψτε στον Γκουίντο Σακόνη να παρουσιάσει ε, το θέμα του με ησυχία σας παρακαλώ. Γκουίντο, έχεις το λόγο. Ευχαριστώ είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό γιατί με αυτή την τροπολογία που πήραμε, την πρωτοβουλία που πήραμε, ε, μπορούμε να παίξουμε άξια τον ε, ρόλο μας, ε, δηλαδή να είμαστε πραγματικά οι φύλακες και οι επιτηρητές της καλής εφαρμογής του Ρίτσο. Ξέρετε ότι τον Φεβρουάριο η Επιτροπή παρουσίασε στα πλαίσια της Επιτροπολογίας μία έκθεση σε σχέση με τον τρόπο εφαρμογής του Ρίτσο ε, και πρόκειται ε, για, το για ένα παράρτημα στην προηγούμενη ε, οδηγία 76-79 και τελικά πρόκειται για, τις, για τους διάφορους περιορισμούς οι οποίοι υπάρχουν στην αγορά σχετικά με τις επικίνδυνες ουσίες. Με την απόφαση αυτή η Επιτροπή ε, ανάμεσα σε άλλες επικίνδυνες ουσίες όπου βεβαίως υπάρχουν ε, περιορισμοί ως προς την αδειοδότηση υπάρχει μια ρύθμιση ε, σχετικά με τις ίνες αμοιάντου, ίνες αμοιάντου οι οποίες είναι διαζώντως επικίνδυνες. Λοιπόν, μέσα σε, σε αυτό το πλαίσιο άλλη μια φορά επιβεβαιώνεται η δυνατότητα να υπάρξει μια μεταβατική περίοδος για ορισμένες χώρες μέλη. Ε, αυτό βέβαια κάτω από πολύ συγκεκριμένους, με πολύ συγκεκριμένους όρους ε, σχετικά δηλαδή με αυτές τις ίνες αμοιάν. Ορισμένες χώρες ζήτησαν μια παράταση, μια μεταβατική περίοδο. Και βεβαίως αυτό αναφέρεται και σε ορισμένα άρθρα τα οποία αφορούν ε, στις Σίνες Αμιάντου. Ξέρετε βεβαίως ότι ε, μέχρι το 2011 έχουμε, μια, έχουμε την προθεσμία για την πλήρη εφαρμογή του, προεγω, του προγράμματος REACH ε, και βεβαίως προσπαθήσαμε να ετοιμάσουμε με τη συνεργασία βεβαίως ε, των άλλων πολιτικών ομάδων μια πρόταση. Ε, αυτό που θέλουμε είναι να ζητήσουμε από την ε, Επιτροπή να υπάρξει μια αυστηρότητα γιατί θα πρέπει μέχρι το 2015 να υπάρχει μια γενική εφαρμογή των διατάξεων του ΡΙΤΣ. Λοιπόν, και βεβαίως ε, θα πρέπει να είμαστε όπως είπαμε πολύ αυστηροί σε οποιασδήποτε παρεκκλήσεις ε, μετά, δηλαδή δεν θα υπάρχει καμία παράκληση μετά από το 2015. Ε, και ακριβώς γι' αυτό θα πρέπει να εκπονήσουμε μια στρατηγική για τον τρόπο που θα διαχειριστούμε τις εφαρμογές αυτών των διατάξεων. Ε, και βεβαίως υπάρχει το θέμα της ε, καταστροφής ε, και της απομάκρυνσης των ινών του αμοιάντου όπου αυτές υφίστανται αυτή τη στιγμή. Ξέρετε πόσο επικίνδυνος είναι ο αμοιάντος, ξέρετε ότι υπάρχει ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα και βεβαίως γι' αυτό το λόγο κάθε παρέκκληση πρέπει να κρίνεται με πολύ μεγάλη αυστηρότητα. Αυτά. Ευχαριστούμε πολύ. Γκουίντο. Λοιπόν, ο Τζον Μπόουις, σαν σκιώδης εισηγητής, «Δακόρντο» λέει ο κύριος Μπόουις. «Δακόρντο», «Δακόρντο», αυτό είπε. Συμφωνεί δηλαδή. Σημαίνει ότι είστε υπέρ, ότι δεν υπάρχει καμία διαφωνία, δεν υπάρχει καμία αντίρρηση. Ναι, ε, ε, θα ήθελα να χρησιμοποιήσω λίγο περισσότερο χρόνο από τον ε, φίλο μου τον Τζον Μπόις γιατί έλαβα μέρος σε μια συνάντηση που αναφερόταν στον αμίαντο. Ε, ξέρετε ότι υπήρχε έκθεση στον αμίαντο για πολλά χρόνια και ξέρετε ότι υπήρχαν πάρα πολλά θύματα από τον αμίαντο και βεβαίως ζητήθηκε ε, και μια παρέκκληση από ορισμένους μέχρι το 2018. Λοιπόν, η έκθεση στον αμίαντο ήταν πάρα πάρα πολύ ε, επικίνδυνη ε, και είναι κάτι το οποίο εμένα προσωπικά με πλήττει, δηλαδή οποιαδήποτε παρέκκληση με, με πειράζει προσωπικά και πραγματικά έχουμε μια ψηφοφορία η οποία αναφέρεται σε πολύ συγκεκριμένες ημερομηνίες γιατί πρέπει τελικά να ξεφύγουμε από αυτόν τον εφιάλτη. Πρόκειται για ένα πραγματικό εφιάλτη ο οποίος έπληξε τις ζωές χιλιάδων ανθρώπων. Λοιπόν, έχουμε... Έναν, ε, έχουμε μια ευθύνη, έχουμε μια ευθύνη ηθικού χαρακτήρα, δεν μπορούμε να δεχθούμε παρεκκλήσεις σε σχέση με τον αμίαντο, ε, χωρίς ε, να λάβουμε υπόψη μας ε, το ηθικό βάρος. Λοιπόν, σας παρακαλώ πάρα πολύ να ληφθεί υπόψη ότι χάθηκαν ανθρώπινες ζωές. Ευχαριστώ. Ναι, ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. εκπλήσωμαι γιατί αυτή η συζήτηση φαίνεται να διεξάγεται μεταξύ Ιταλών αυτή τη στιγμή αλλά εγώ προσωπικά θα ήθελα να υπογραμμίσω τις ε, πτυχές ε, οι οποίες ε, δεν αφορούν μόνον το θέμα της, του γαμιάντου γιατί είναι ένα θέμα που δεν αφορά μόνο τα πρόσωπα τα οποία έχουν εκτεθεί Πρόκειται επίσης για άλλα άτομα τα οποία τελικά καθάριζαν και είχαν και αυτά εκτεθεί είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ ε, σημαντικό. Πρέπει να καταλάβουμε την σοβαρότητα του ζητήματος και πρέπει πραγματικά να καταλήξουμε σε μία λύση η οποία θα εφαρμοστεί μακροπρόθεσμα. Γιατί πρόκειται τελικά ε, για, για την αποσύνθεση του ε, δηλαδή για την ε, δυνατότητα που έχουν οι ίνες του αμοιάντου να εισέλθουν στο αναπνευστικό σύστημα. Και πραγματικά δια της εισπνοής ε, υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλοι κίνδυνοι ε, και πρέπει να καταλάβουμε ότι η εισπνοή του αμοιάντου είναι κάτι το πάρα πολύ επικίνδυνο και βεβαίως πρόκειται για ίνες οι οποίες μπορούν τελικά μέσω του αναπνευστικού συστήματος ε, να εισέλθουν στον οργανισμό και πρέπει τελικά να καταλάβουμε ότι πρόκειται για ένα πάρα πάρα πολύ ε, σημαντικό πρόβλημα πρέπει να κάνουμε κάτι, πρέπει να υπάρξει μια πραγματική απομάκρυνση ε, αυτών των υλικών μέσω της απορρόφησής τους και της ιαλοποίησής τους. Ευχαριστώ, ο Καλ Σλούτα. Ευχαριστώ, ε, κύριε Πρόεδρε. Ε, πιστεύω ότι υπάρχει ένα μικρό πρόβλημα. Ε, πότε επιτέλους ε, θα έχουμε ε, ένα, μια ρύθμιση σε σχέση με τα απόβλητα, με τα απόβλητα του αμοιάντου. Είναι κάτι το οποίο μας το υποσχεθήκατε και ακόμα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Δεν... Δεν βλέπω κανέναν άλλον, οπότε θέλω να ακούσω τον εκπρόσωπο της Επιτροπής, ο κύριος Κλωσ Μπέρεντ. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Σακώνη πρώτα απ' όλα για τη δουλειά που έκανε, για την αναθεώρηση του σχέδιου κανονισμού και για το ψήφισμα που προετοίμασε και σας διαβεβαιώ ότι ουδέποτε είχαμε πρόθεση να πισχνάσουμε τις ε, διατάξεις και τους περιορισμούς για τον αμίαντο σε καμία περίπτωση και φυσικά θέλουμε και εμείς όπως και το Κοινοβούλιο ε, ολική κατάργηση.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 Μιλάμε για τους περιορισμούς για όλες τις ουσίες ε, που εγκρίθηκαν τα τελευταία 30, 30 χρόνια ε, στο παράρτημα 9 του ΡΙΤΣ και στον 76-79 και ε, τα κράτη-μέλη θα πρέπει να προσαρμοστούν στο νέο νομικό περιβάλλον ώστε να εφαρμοστούν καλύτερα οι διατάξεις και να είναι σαφέστερες. η παρέκκληση που, στην οποία αναφέρθηκε τώρα ο κύριος Σακονή για τα διαφράγματα και τους ηλεκτρολίτες υπήρχε ήδη στην κείμενη νομοθεσία. Τέσσερα κράτη-μέλη χρησιμοποιούν αυτή τη διάταξη. Το 2006-2007 έγινε αναθεώρηση. Αποκινούμε τα κράτη-μέλη και τι ενδιαφερόμενε επιχειρήσει και τελικά μα έστειλαν τα σχόλιά του για αυτέ τι εξαιρέσει. Ο κανόνα που έχετε λοιπόν ε, δεν ε, αποδυναμώνει τι διατάξει σε καμία περίπτωση. Η επόμενη αναθεώρηση προβλέπεται για το 2011 διότι ξέρουμε ότι ε, συνεχίζουν οι επιχειρήσει να προσπαθούν να βρουν ουσίε προ αντικατάσταση και θα ολοκληρωθούν οι εργασίες γύρω στο 2011. Επίσης, ο χειρισμός των αποβλήτων που ανέφερε ο κύριος Πρόεδρος στη δήλωσή του μας απασχολεί και πήραμε πληροφορίες από τις επιχειρήσεις ε, και ούτως ή άλλως οι ίνες ε, ε, μετατρέπονται σε ίνες γυαλιού και δεν έχουν καμία σχέση πλέον με τον αμίαντο μετατρέπονται, δηλαδή όποτε δεν υπάρχουν απόβλητα. Θα έρθω σε επαφή με τους συναδέλφους μου από τη ΓΑΜΑ Περιβάλλον για τα υπόλοιπα. Δεν μπορώ να σας απαντήσω τώρα, διότι δεν είναι αρμοδιότητα της δικής μου υπηρεσίας, αλλά ε, θα απαντήσουν οι συνάδελφοι από τη ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ Ευχαριστώ. Μπορούμε να ψηφίσουμε για την προφορική ερώτηση και το σχέδιο ψηφίσματος. Α, όχι. Ο κύριος Σακώνη θέλει πάλι το λόγο. Παρακαλώ. Ναι. Θέλω μόνο να υπογραμμίσω μία πτυχή, ένα θέμα ε, το οποίο δεν το, το αντιπαρήλθα. Ε, δεν συμφωνήσαμε να δεχθούμε αυτές τις ε, αναβολές Πρόκειται για τέσσερις ευρωπαϊκές χώρες οι οποίες ζήτησαν μια παράταση, αλλά δεν πρόκειται μόνο για αυτή την παράταση. Ε, πρόκειται απλά και μόνο για την ερμηνεία ορισμένων άρθρων και για τις ε, διατάξεις που αναφέρονται ε, στην αγορά για τον μέχρι το 2015. Αλλά προσοχή, υπάρχει ένα πρόβλημα. Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι στην Ευρώπη διαχειριζόμαστε καλά αυτό το πρόβλημα, δηλαδή σε σχέση με αυτό το πάρα πολύ επικίνδυνο υλικό. Υπάρχει το θέμα των χωρών παραγωγών αυτής της πολύ επικίνδυνης ουσίας και βεβαίως αυτό είναι ένα ηθικό πρόβλημα. Έχουμε μεγάλη ευθύνη, το ξέρω και θα ήθελα πολύ απλά να το υπογραμμίσω και να πω ότι πρόκειται ε, για μια τεχνική πτυχή. Ε, υπάρχουν ορισμένα λάθη. Θέλετε να να αναφερθώ σε αυτά τα λάθη που υπάρχουν. Ε, δεν ξέρω. Υπάρχουν δύο-τρία λόγια τα οποία θα πρέπει να τα. δύο-τρει λέξει οι οποίε θα πρέπει να διαγραφούν. Περί αυτού πρόκειται. Δηλαδή πρόκειται για τη λεκτική διατύπωση. Θέλετε να νομίζω ότι αν μπορεί να υπάρξει μια λύση σε επίπεδο επιτροπής, αυτή η λύση πρέπει να δοθεί σήμερα. Λοιπόν, κατάλαβα τι ζητήσατε. Μπορείτε να το εξηγήσετε τώρα. Λοιπόν, πρόκειται για μερικές τροποποίησεις, έτσι. Ο Τζον. Επιβεβαιώνω αυτά που είπε ο κύριος Σακώνη, ότι όλοι λάβαμε αυτές τις μικρές αλλαγές που έγιναν, συμφωνούμε όλοι, οπότε ας ψηφίσουμε για το σύνολο. Ωραία. Άρα δεν χρειάζεται να κάνουμε λοιπές δηλώσεις. Όλοι έχουν ενημερωθεί, οι πολιτικές ομάδες έχουν πάρει τις προτάσεις, τις ε, ε, τροπολογίες ίσων σημασίας. Θα ψηφίσουμε για την προφορική ερώτηση και μετά θα ψηφίσουμε για το σχέδιο ψηφίσματος. Είναι όλα σαφή για σας, πολύ ωραία. Ηλεκτρονική ψηφοφορία πρώτα απ' όλα ή γίνεται χωρίς Ποιοι είναι υπέρ. Υπέρ της προφορικής ερώτησης παρακαλώ με ένα τεσχυρός κατά αποχές εγκρίθηκε σαφέστατα. Και ποιοι είναι υπέρ του σχεδίου ψηφίσματος όπως τροποποιήθηκε. Χρειαζόμαστε ονόματα ηλεκτρονικά. Λοιπόν, παρακαλώ. Ο Ανδρέας προτείνει ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ψηφίστε παρακαλώ. Ψηφίσατε. Πέρας. 16 υπέρ, κανείς κατά, τέσσερις αποχές. Ευχαριστώ και συγχαρητήρια κύριε Σακών. Να σας πω απλά ότι στην Ολομέλεια προς το παρόν έχει προβλεφθεί για ε, το δεύτερο ήμιση του Απριλίου ή Μάιο. 15, ε, το επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης, εκθεσή της Επιτροπής Περιβάλλοντος ε, για τον απολογισμό της Αντιπροσωπείας Επιτροπής στην Κωνσταντινούπολη. Θέλω να δώσω το λόγο στους ε, όσους μετήχαν σε αυτή την αντιπροσωπεία για να φράσουν την άποψή τους. Κριστίνα Γκουτιέρες Κορτίνες, ε, επικεφαλής της αντιπροσωπείας. Θέλετε το λόγο, θέλετε. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Νομίζω ότι είναι ένα θέμα ε, στο οποίο δόθηκε πολύ μεγάλη ε, δημοσιότητα. Ακούστηκαν πολλά πράγματα στον τύπο σχετικά με αυτό το φόρουμ αλλά εγώ διαρωτώ με τελικά σε τι χρησιμεύσε αυτό το φόρουμ, ποιοι ήταν οι στόχοι που είχε θέσει και αν τελικά πραγματοποιήθηκαν οι στόχοι αυτοί. Ξέρετε ότι έχουμε την UNESCO ε, στα παρασκήνια ε, και το ΝΑΤΟ τελικά θέλουμε να βελτιώσουμε τις δυνατότητες πρόσβασης στο νερό σε όλες τις κοινωνίες, για όλες τις ε, χώρες, για όλες τις κοινωνίες. Και βεβαίως θα πρέπει να υπάρξει και μια ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των χωρών για να δούμε ποιες είναι οι δυνατότητες που υφίστανται αυτή τη στιγμή. Το ζήτημα αποτίθεται είναι πού βρίσκονται οι υπουργοί. Τι κάνουν οι υπουργοί αυτή τη στιγμή, γιατί τελικά πρόκειται για υπουργικέ αποφάσεις. Τελευταία ανάλυση οι υπουργοί αποφασίζουν. Έχουμε λοιπόν ένα ψήφισμα ε, το οποίο εκπονήσαμε ε, και θέλουμε το νερό να θεωρηθεί ένα θεμελιώδες δικαίωμα. Και τι είπαν τελικά οι δημοσιογράφοι. Οι δημοσιογράφοι είπαν ότι απέτυχε αυτό το φόρουμ γιατί αυτό το αξίωμα ε, δεν έγινε αποδεκτό. Ε, θα ήθελα λοιπόν να λάβετε υπόψη τις δικές μου απόψεις. Υπάρχουν μόνο 19 χώρες οι οποίες υποστηρίζουν ότι είναι ανθρώπινο δικαίωμα. Ε, ξέρετε ότι το, ο Καναδάς είναι μια χώρα η οποία είναι κατά της άποψης αυτής. Λοιπόν, διερωτόμαστε γιατί ο Καναδάς να είναι κατά αυτής της άποψης, κατά αυτής της ιδέας. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι αν έχουμε σαν μοναδικό στόχο να περιληφθεί στα ανθρώπινα δικαιώματα η πρόσβαση στο νερό ε, πρόκειται για μια αποτυχία αυτού του φόρουμ. Αλλά δεν έχουμε μόνο αυτό το στόχο, έχουμε μια σειρά στόχων. Ε, υπάρχουν εξαιρετικά ψηφίσματα τα οποία εγκρίθηκαν από το Κοινοβούλιο. Αλλά πρέπει να δούμε γιατί υπάρχει τόση αντίσταση, τόση αντίρρηση. Ε, γιατί, γιατί δεν γίνεται δεχτή αυτή η αρχή. Ίσως δεν αναπτύξαμε αρκετά αυτή την αρχή. Ο Καναδάς θεωρεί ότι αν πρόσβαση σε νερό ποιότητας αποτελεί ένα ανθρώπινο δικαίωμα, εάν υπάρξει παραδείγματο χάρη μια πλημμύρα και το νερό δεν είναι πια πόσιμο, ε, τι θα γίνει, τι θα κάνουμε. Ε, υπάρχει το θέμα τις ευθύνες Δεν μπορέσαμε μέχρι στιγμής ε, να θέσουμε ε, τις προϋποθέσεις για το ποιος φέρει την ευθύνη. Υπάρχουν πολλές χώρες τις οποίες οι κυβερνήσεις δεν εγγυώνται ε, ότι το νερό είναι πόσιμο. Προέρχομαι από τη βόρεια ε, Ισπανία. Λοιπόν, όταν έχουμε πλημμύρες, το νερό δεν είναι πια πόσιμο, ε, γιατί δεν έχουμε τη δυνατότητα, δεν υπάρχουν οι απαραίτητες εγκαταστάσεις για τον καθαρισμό του νερού. Ε, και θα πρέπει λοιπόν να καταλάβουμε και να δούμε τι εννοούμε όταν λέμε ότι το νερό, η πρόσβαση στο νερό είναι ένα θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα. Πρέπει να ξέρετε ότι όλοι στο Κοινοβούλιο υποστηρίξαμε και πρόκειται για ένα κοινό στόχο ότι τα δικαιώματα του ανθρώπου ε, δεν ε, είναι κάτι το αφηρημένο. Είναι κάτι για το οποίο θα πρέπει να δεσμευτούν όλες οι χώρες, γιατί διαφορετικά δεν υφίστανται ανθρώπινα δικαιώματα. Πρέπει οι χώρες μέλη να δεσμευτούν και θα πρέπει πραγματικά να επιτρέψουν στους πολίτες την προστασία η οποία είναι αναγκαία για να πραγματοποιηθούν, για να έχουν σάρκα και οστά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Λοιπόν, θα πρέπει αυτό το ανθρώπινο δικαίωμα ε, να μπορεί να είναι σεβαστό σε όλες τις χώρες μέλη. Θα πρέπει να κάνουμε ορισμένες αναλύσεις. Υπάρχει μια νομοθετική πτυχή. Υπάρχει ε, επίσης ε, το θέμα της επιβολής ε, κυρώσεων. Τι γίνεται όταν έχουμε ποταμούς οι οποίοι τελικά είναι μολυσμένοι. Τι θα κάνουμε. Θα πρέπει να υπάρξουν νομοθετικά κείμενα, ποιοτικά νομοθετικά κείμενα, τα οποία θα πρέπει να εφαρμόζονται όχι μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά σε όλη την Ευρώπη. Λοιπόν, όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά. Αλλά υπάρχουν και άλλα ζητήματα, υπάρχουν και άλλα θέματα, τα οποία κατά τη γνώμη μου είναι πάρα πολύ σημαντικά. Πάντως κάτι άρχισε να κινείται αυτή τη στιγμή. Έχουμε ε, μια πολύ σημαντική διαφωνία ε, σχετικά με τα διασυνοριακά ύδατα. 60% των υδάτων του πλανήτη προέρχεται από ποταμούς οι οποίοι περνάνε τα σύνορα εντό εισαγωγικών και βεβαίως ε, είναι πάρα πολύ δύσκολο να δούμε ποιος έχει την ευθύνη και στην Ισπανία έχουμε πάρα πολλά ε, προβλήματα Έχουμε ορισμένες ε, συμφωνίες ε, με την Πορτογαλία, υπάρχει μια συμφωνία η οποία υφίσταται ώστε να υπάρξει ένας επιμερισμός των ευθυνών σχετικά με την ποιότητα των υδάτων. Αλλά καταλάβαμε ότι οι Τούρκοι αυτή τη στιγμή έχουν άλλα προβλήματα. Έχουν πρόβλημα με την ε, Συρία και δεν ήμασταν αρκετά προσεκτικοί ε, τελειώνω, τελειώνω, αμέσω τελειώνω. Ε, ποιο ήταν το άλλο θέμα το οποίο ε, εξετάστηκε. Υπήρξε μία ε, συνεδρίαση η οποία αναφερόταν στις εργασίες της UNESCO. Εδώ πραγματικά έγινε μια εξαιρετική δουλειά ώστε να μπορούμε να έχουμε την διάγνωση των προβλημάτων Βεβαίως υπάρχει έλλειψη υποδομών, υπάρχει έλλειψη εκπαίδευσης, ε, κατάρτισης, νομοθεσίας και βεβαίως υπάρχει και έλλειψη χρημάτων. Ανάγκη στη χρημάτων επί του θέματος. Λοιπόν, μείναμε πάρα πολύ ε, και ε, υπάρχει αυτό το πρόβλημα μεταξύ των υδάτων δημόσιου και ιδιωτικού χαρακτήρα και υπάρχει ένα ψήφισμα σύμφωνα με το οποίο είπαμε ότι θα πρέπει να υπάρξει μια ισορροπία μεταξύ του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα. Θα πρέπει να ασκείται ένας έλεγχος, θα πρέπει να υπάρχει ένα σύστημα επιτήρησης ε, για τον ιδιωτικό τομέα και είναι κάτι το οποίο θα πρέπει ε, να το προσέξουμε πάρα πολύ. Ίσως ο συνάδελφος θα πρέπει να πάρει το λόγο. Είναι ένα θέμα συνδικαλιστικό επίσης. Θα πρέπει βέβαια να λάβουμε υπόψη αυτό που λένε τα συνδικάτα ότι θα πρέπει να έχει δημόσιο χαρακτήρα αυτή η επιτήρηση. Και υπάρχει και άλλο ένα σημείο το οποίο είναι πραγματικά σημαντικό και όπου δυσκολευτήκαμε να επιτύχουμε μια συμφωνία, δεν συμφωνήσαμε εμείς κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι μεταξύ μας, πρόκειται για την ε, αρχή της αλληλεγγύης σχετικά με την διάθεση του ύδατος, με τον επιμερισμό των ευθυνών και αυτό είναι το βασικό πρόβλημα. Και στην Αφρική και στη Μέση Ανατολή υπάρχουν χώρες ε, από τις οποίες περνάνε ποτάμια. Ε, η Γάζα, ας πούμε, η Συρία θα πρέπει να μοιραστεί το νερό και να συμφωνήσει με το Ισραήλ. Επαναλαμβάνω, δεν είναι εθνικά θέματα. Τα ποτάμια δεν ξέρουν, δεν γνωρίζουν σύνορα. Και είναι θέμα το ΟΗΕ και από την αρχή αυτό λέμε. Τελικά πιστεύω τα πράγματα κινήθηκαν. Βλέπουμε ότι υπάρχουν περισσότερες χώρες που προσπαθούν να έχουν ε, έλεγχο στην ποιότητα των υδάτων. Τονίζεται πολύ ο ρόλος των γυναικών, αλλά τώρα δεν το βλέπω. Δεν βλέπω ότι γίνεται στο Μεξικό. Βέβαια, Υπάρχουν μεγάλα προβλήματα οικονομικά και πολλοί είναι απόντες από αυτή τη συνάντηση του Μεξικού. Θα δω τι θα πούν και οι συνάδελφοι, αλλά θα πρέπει να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για να θεωρείται δικαίωμα το νερό που διατίθεται. Και να κοιτάξει η Ευρώπη τι θα κάνει με αυτούς που παραβιάζουν αυτό το ανθρώπινο δικαίωμα. Για να ξέρουν οι χώρες που προσυπογράφουν σε τι δεσμεύονται. Ευχαριστώ πολύ. Uh, Σας ευχαριστούμε. Ο κύριος ε, Μουσάκιο, έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ. Η Κριστίνα είπε πολλά και τα είπε πολύ καλά θα ήθελα να την ε, ευχαριστήσω γιατί ήταν αυτή που ήταν η πρόεδρος της Επιτροπής μας, έκανε πολύ καλή δουλειά ε, και βεβαίως μπορούμε να κάνουμε, ε, υπάρχει ένα, μια έκθεση, ένα είδος ρεπορτάζ για τις εργασίες μας. Θα ήθελα να το συστήσω στους συναδέλφους, υπήρξε εκπροσώπηση πολλών χωρών και επίσης της κοινωνίας Υπήρξαν 55 πολίτες ε, οι οποίοι ήρθαν από την Ιταλία και οι οποίοι έλαβαν μέρος σε αυτό το φόρουμ. Ε, υπήρξε επομένως μια κοινωνική ευρύτατη εκπροσώπηση. Δουλέψαμε καλά. Θα ήθελα να πω ε, και η Κριστίνα αναφέρθηκε σε αυτό στην αρχή ότι τα τελικά αποτελέσματα δεν έγιναν αποδεκτά με ικανοποίηση και στον Ιταλικό τύπο. Γιατί δεν καταφέρουμε τελικά να αναγνωρίσουμε το νερό σαν ένα θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα. Ε, και βεβαίως ε, δεν καταλήξαν ούτε 29 χώρες ε, και αυτοί που διαφώνησαν είπαν ότι αν αναγνωρίσουμε ότι είναι θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα το νερό, τότε θα πρέπει αυτό που θα πούμε να, μπορούμε, να είμαστε και σε θέση να το πραγματοποιήσουμε. Ε, γιατί είπαμε ότι αυτό το ε, φόρουμ είχε έναν ελεύθερο χαρακτήρα ε, και βεβαίως το γεγονός του ότι υπήρχε μια συμμετοχή της UNESCO και του ΝΑΤΟ ε, δεν σημαίνει ότι μπορούσαμε και να καταλήξουμε. Το 1992 είχαμε μία ε, διάσκεψη για το μέλλον της γης και τελικά καταλήξαμε ε, στην βιοπικιλότητα, ε, καταλήξαμε σε, στην προστασία του περιβάλλοντος, αλλά δεν μπορέσαμε να καταλήξουμε στην αναγνώριση του δικαιώματος του νερού σαν ένα ανθρώπινο δικαίωμα. Γιατί υπάρχουν όχι μόνο ιδιωτικά ε, συμφέροντα, αλλά υπάρχουν και άλλες ε, συνθήκες. Ε, έχουμε μία συνθήκη αυτή τη στιγμή για, το κλίμα. Έχουμε το πρωτόκολλο του Κιώτο, υπάρχει μία δέσμευση μετά από αυτή τη συνθήκη. Εδώ δεν καταλήξαμε σε, σε τίποτα το δεσμευτικό, δεν υπάρχει καμία δεσμευτική συνθήκη. Άκουσα αυτά που είπε η Κριστίνα και πιστεύω ότι όπως γράψαμε στο κείμενο αυτό. Ε, όλα αυτά, το είπαμε και στην Κοπενχάγη, ε, το, οι αλλαγές του κλίματος επηρεάζουν άμεσα την ποιότητα του νερού. Λοιπόν, πρέπει ε, να τα δούμε όλα αυτά σε μια αλληλεξάρτηση, δηλαδή την αλλαγή του κλίματος με την αλλαγή ε, της ποιότητας του νερού. Κατά τη γνώμη μου θα πρέπει να υπάρξει ένα πρωτόκολλο για το νερό ένα πρωτόκολλο το οποίο θα έχει δεσμευτικό χαρακτήρα έτσι ώστε να μπορούμε να είμαστε λειτουργικοί, έτσι ώστε να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε αυτά για τα οποία θα αποφασίσουμε. Λοιπόν, και έτσι μπορούμε και να δεσμευτούμε και ως προς τους πολίτες, ε, διότι εδώ θέλουμε να υπάρξει αναγνώριση του νερού σαν ένα βασικό ανθρώπινο δικαίωμα. Είναι, Μπορεί να αναγνωρίσει ο καθένας ότι το νερό είναι είδος πρώτης ανάγκης. Λοιπόν, νομίζω ότι μπορούμε να προχωρήσουμε και να κερδίσουμε μία μάχη σε αυτό τον πόλεμο. Τα είπε όλα αυτά πολύ καλά η Κριστίνα. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, άλλο ε, με, μέλος της αποστολής ήταν η κυρία Σάντα. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Και εγώ θα ήθελα να παρέμβω και να πω πολύ απλά ε, λίγα πράγματα παραπάνω σε σχέση με τα όσα είπαν ε, οι συνάδελφοι. Πιστεύω ότι ε, ήταν πολύ σημαντική η συμμετοχή μας. Είχαμε διμερείς επαφές που ήταν πάρα πολύ σημαντικές και πρέπει να πούμε ότι ε, υπήρξε μία συνεννόηση και συμφωνία ε, μεταξύ όλων αυτών που έλαβαν μέρος σε αυτό το συνέδριο. Εμείς ε, θέλαμε να υπάρχει ένα ψήφισμα. Εμείς τελικά συμφωνήσαμε με το ψήφισμα του, του Κοινοβουλίου για να μπορέσουμε να αγωνιστούμε και να προσπίσουμε το, το νερό σαν ένα θεμελιώδες δικαίωμα και στην Υπουργική Διάσκεψη είχαμε ε, την ίδια θέση αλλά και στο Κοινοβούλιο, στην Κοινοβουλευτική Διάσταση το ίδιο. Φαίνεται λοιπόν στη ψηφοφορία, στη δεύτερη ημέρα, ότι αυτό μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Και το δικαίωμα πρόσβαση στο νερό, όχι μόνο το νερό αυτό καθευτό, σε εξυγίανση του νερού, γιατί είναι δημόσιο αγαθό και θα πρέπει να διατηρείται σε δημόσιο έλεγχο το νερό. Και μια σειρά μέτρων προτείναμε για να αυξηθούν οι πόροι που διατίθεται εκεί, τα χρήματα. Και κάποια στιγμή για την επόμενη θητεία ίσως θα μπορούσε να είναι ε, μια υπόθεση για τους εκπροσώπους και του ΙΕ και της UNESCO για το υδρολογικό πρόγραμμα, για το νερό γενικότερα. Αυτό που καταλάβαμε λοιπόν ήταν ότι χρειάζεται να περάσουμε σε ένα μελλοντικό πλαίσιο τέτοιου είδους παγκοσμίων φόρων ε, ε, τέτοια φόρα να έχουμε δηλαδή και όχι εθνικά. Ε, όταν καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει ένα πρόβλημα με το νερό, ακόμα συνηθίζουμε να λειτουργούμε σε ιδιωτικό πλαίσιο, ε, με διαφόρους ενδιαφερόμενους και τα λοιπά, αλλά θα ήταν καλύτερο αυτό να το βλέπουμε διεθνώς. Είναι παγκόσμια συζήτηση, είναι παγκόσμιο το θέμα. Στον ΟΗΕ δηλαδή. Και όπως έλεγε το ψήφισμά μας, θα πρέπει να συνδέεται η πρόσβαση ε, στο νερό και η εξηγίασή του και για το πακέτο της κλιματικής αλλαγής το υποστηρίξαμε και τα κοινοβούλια και της Λατινικής Αμερικής και της ε, Αφρικής. Το είδα πάρα πολύ θετικά αυτό, να ενισχυθεί ο ρόλος δηλαδή του δικαιώματος αυτού στο νερό και στο καθαρό νερό για τη μετά και ότο εποχή και μετά την Κοπεχάγη. Αυτά. Είχαμε επαφές και με τα συνδικάτα και θα ήθελα να σας θυμίσω ότι υπάρχει ένα αίτημα σημαντικό. Η οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση επηρεάζει πάρα πολύ έντονα και αποφασιστικά τις εταιρείε που ιδιωτικοποίησαν εδώ και καιρό την πρόσβαση στο είδωρ. Η Βρετανία, ας πούμε, πριν από 20 χρόνια. Ήταν ισχυτικό το παράδειγμα αυτό. Και οι εργαζόμενοι ζήτησαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εμβαθύνουμε εκεί, να εξετάσουμε τη βιωσιμότητα σε περιόδους κρίσεως που είναι πάρα πολύ επισφαλής η κατάσταση και πάρα πολύ ε, συγκρουσιακή. Για να μην είναι τελείως ιδιωτικοποιημένη η υπόθεση της διαχείρισης των υδάτων στα χέρια ιδιωτών, δηλαδή γιατί σε περίοδους κρίσεων βλέπουμε τι γίνεται. Αυτά από πλευράς αντιπροσωπείας. Και επαναλαμβάνω ήταν πολύ ενδιαφέροντα όλα και ευχαριστώ τη γραμματεία που μας διευκόλυνε. Ευχαριστώ πολύ. Thank Σας ευχαριστώ. Άλλος κανείς? Όχι. Σας ευχαριστώ πολύ. Την κυρία Κουτιές Κορτίνες, την ε, Ινέσα Γιάλα και τον κύριο Μουσάκιο που μας ε, ανέφεραν ε, για τα σημαντικά αυτά που συζήτησαν εκεί στο φόρουμ για το είδο. Και ερχόμαστε τώρα στο τελευταίο μας θέμα. Ορίστε. Ναι, το τελευταίο είναι. Γιατί κάνετε έτσι. Παρουσίαση της ΣΤΟΑ. Η αξιολόγηση επιστημονικών και τεχνικών επιλογών θα μας τα παρουσιάσει αυτά η Ντορέτ Κόρμπεϊ. Παρακαλώ, έχετε το λόγο, κυρία μου. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Σύντομα θα τα πω, δεδομένου και του ακροτηρίου. Και στην Είναι η τελευταία συνεδρία της Επιτροπής Περιβάλλοντος. Οι συνάδελφοι που συμμετείχαν στις ε, προηγούμενες ηττίε συνδέουν τη στοά με τα σοκολατούχα αυγά κίντερ αυτά και τα διάφορα παιχνίδια που βρίσκει κανείς μέσα. Πριν από δυόμιση χρόνια. Και πραγματικά πρέπει να σας πω ότι έχει παρέλθει αυτός ο καιρός της έκπληξης των αυγών κίντερ. Είχε γίνει μεγάλη φασαρία τότε. Ήταν πολύ ε, επιτυχημένα τα προγράμματα που ξεκίνησαν και για μας, για το περιβάλλον, τη δημόσια υγεία και την ασφάλεια των τροφίμων. Σύντομα, να σας αναφέρω, δεν έχει νόημα τώρα να μπούμε ε, σε λεπτομέρειες όλων των σχεδίων και όλων των έργων, αλλά καλό θα ήταν να τα παρακολουθήσετε όλοι και να σας ενημερώσω ότι σε μερικές εκθέσεις της ΣΟΑ αναφέρονται διάφορα πράγματα. Πλήρης περιγραφή των προγραμμάτων ε, περιλαμβάνεται στην ετήσια έκθεση της ΣΤΟΑ. Κανονικά την έχετε λάβει όλοι στα έδρανά σας. Πάρα πολύ σύντομα να πω δύο λόγια. Έχουν γίνει πολύ ε, σημαντικές μελέτες τα τελευταία χρόνια. Πρώτον, ε, τεχνολογίες... Ε, του μέλλοντος είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Είναι, είναι συναρπαστικό να δούμε τι γίνεται με τη γενετική τεχνολογία, τη βιοτεχνολογία και τη τεχνολογία ηλεκτρονικών υπολογιστών όταν συγκεντρώνονται όλα αυτά. Τι σημαίνει για τον άνθρωπο και για την κοινωνία. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα και η έκθεση και η συζήτηση που έγινε. Σας το συνιστώ. Μετά από δυόμιση χρόνια μπορώ πραγματικά να σα συστήσω να το διαβάσετε. Είναι καταπληκτική η έκθεση αυτή πάρα πολύ επίκαιρα και τα συμπεράσματα. Δεύτερον, επίτευγμα της ΣΤΟΑ. Η προβληματική της αντοχής στα αντιβιωτικά. Όλοι εδώ γνωρίζετε ότι η αντοχή στα αντιβιωτικά είναι τεράστιο πρόβλημα. Και σε πολλά κράτη τα δίνουν ε, έτσι χαλαρά και χωρίς κανένα πρόβλημα όχι μόνο στους ανθρώπους αλλά και στα ζώα. Γίνεται άκρα τη χρήση και τη χρήση αντιβιωτικών. Και έτσι αναπτύσσονται μικρόβια που ε, εμφανίζουν αντίσταση στα αντιβιωτικά και είναι πάρα πολύ δύσκολο να καταπολεμηθούν. Και εδώ θέλει προσοχή να το διαβάσετε. Άλλα θέματα που δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμα. Η παγκόσμια δημόσια υγεία, η ατζέντα της έρευνας των φαρμακευτικών εταιριών και τα προγράμματά τους και με ποιο τρόπο μπορούν να έχουν μεγαλύτερη επιρροή οι δημόσιες αρχές για να αντιμετωπίζουν οι φαρμακευτικές εταιρείες καλύτερα τις πραγματικές ασθένειες και τα προβλήματα που υπάρχουν στη δημόσια υγεία. Και θα πρέπει να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε και οι πολιτικοί, τι μπορούν να κάνουν και οι αρχές για να ασχοληθούμε περισσότερο με τα παραμελημένα νοσήματα, neglected diseases λέγονται αυτά. Μελλοντικά συστήματα επίσης ενέργειας, όλοι έχουμε φιλόδοξους στόχους και τους ξέρουμε, 20-20-20, 20% ε, ανανεώσιμες πηγές, 20% μείωση του διοξυδίου του άνθρακα μέχρι το 2020. Πώς μπορούν να γίνουν όλα αυτά. Υπάρχει μελέτη εδώ της ε, ΣΤΟΑ, πολύ ενδιαφέρουσα, Και πολύ ενδιαφέροντα αυτά που μας λέει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Άλλα θέματα που τους απασχόλησαν ήταν οι μεταφορές, πολύ σημαντικό και μεγάλε οι προκλήσει εκεί. Άλλη έκθεση, Human Enhancement. Υπό την αιγίδα της Ρία Όμεν. Τι είναι αυτό. Είναι διάφορες φάσεις για την ενδυνάμωση του ανθρώπου, δεν ξέρω, βελτίωση ε, του ανθρώπου, του ανθρωπίνου σώματος και του ανθρωπίνου πνεύματος. Πώς θα γίνει αυτό. Μπορούν να γίνουν πολλά πράγματα από πλευράς ιατρικής, από πλευράς φαρμάκων και μπαίνουν και διάφορα δεοντολογικά ζητήματα και ηθικά ε, και διάφορες προκλήσεις και τα λοιπά. Έχουμε και άλλα ζητήματα για την ευημερία των ζώων, για την ασφάλεια των τροφίμων, σχέση τροφίμων με δημόσια υγεία, γενετικές δοκιμές και ο ρόλος της τεχνολογίας, της πληροφορία και στις κλιματικές αλλαγές. Αυτά. Πολύ σημαντικά όλα αυτά και επαναλαμβάνω ξανά ότι τα προηγούμενα χρόνια η ΣΤΟΑ έχει κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά και ήταν πραγματικά μεγάλη μου χαρά να συμμετέχω στο πάνελ εκεί. Ήταν πάρα πολύ διδακτικό για μένα και πολύ ενδιαφέρον και πάρα πολύ ψιότητα τη ΣΤΟΑ. Και είναι στρατηγική σημασία οι γνώσει που αποκομίζουμε εκεί και για την Επιτροπή Περιβάλλοντος και για άλλες ε, επιτροπές. Ε, επιθυμίες δεν έχουμε, έχουμε. Η ΣΤΟΑ ακόμα δεν αξιοποιείται ε, όπως θα έπρεπε το θέμα της έρευνας και των μελετών και η σχέση τους με τις ε, κοινοβουλευτικές επιτροπές νομίζω δεν έχει καλυφθεί πλήρως. Εντάξει, συμμετέχουν μέλη όπως εγώ των επιτροπών στο πάνελ της ΣΤΟΑ. Σε εμάς δεν απόκειται να βελτιώσουμε τη σχέση μας, αλλά δεν την αξιοποιούμε όπως θα έπρεπε, όπως θα της άξιζε. Κάναμε διάφορες προτάσεις είναι σημαντικό να δούμε όλες τις εκθέσεις ας για την αντοχή στα αντιβιωτικά και να τις ε, παρουσιάσουμε στις διάφορες επιτροπές. Είχαμε ακροάσεις, κάθε χρόνο γίνεται μια ακρόαση και έρχονται ε, επιστήμονες πάρα πολύ υψηλού επίπεδου αλλά χαμηλή η προσέλευση των μελών του Κοινοβουλίου. Κρίμα, αυτό θα μπορούσε να βελτιωθεί στο επόμενο διάστημα. Αυτά. Δεν έχω τίποτα άλλο να πω. Ήταν η τελευταία φορά που πέρα το λόγο στην Επιτροπή Περιβάλλοντος. Ευχαριστώ κύριο στον Πρόεδρο για τα τελευταία δυόμιση χρόνια και τους συναδέλφους για τη συνεργασία. Αυτά. Τώρα να δούμε τι παρατηρήσεις έχετε και τη σχόλια για την εργασία του πάνελ της ΤΟΣ. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, ήταν και το τελευταίο θέμα. Δεν έχουμε τίποτα στα διάφορα και έχουμε απομείνει πολύ λίγοι. Θα ήθελα να σας δώσω την ευκαιρία τώρα αν θέλετε να κάνετε κάποια προσωπική δήλωση, να βγάλετε κάτι από μέσα σας στην Επιτροπή να πείτε στους πολίτες της Ευρώπης, όποιος θέλει. Μη σπρώχνεστε. Ο Γκουίντο σακώνει. Πες τίποτα για τους πολίτες της Ευρώπης, ακούνε. Αντρές μη. It's, δεν θέλω να σας βασανίσω, ούτε να σας ταλαιπωρώ. Αλλά επειδή έχουμε χρόνο σήμερα, περίεργος, ε, ε, έχουμε εργαστεί σκληρά όλο αυτό το διάστημα. Τώρα που έχουμε λίγο χρόνο, κατ' εξαίρεση, σας δίνω την ευκαιρία να πείτε ό,τι θέλετε. Να κάνετε κάποια δήλωση για να μπει και στο αρχείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σε επιτροπής μας. Καλά. Ε, ο Τζον Μπόις τότε. Πρόεδρε. Φτάνουμε τώρα στη λήξη της επίσημης συνεδρίασης. Είναι ευκαιρία να διαπιστώσουμε ότι και να σημειώσουμε ότι τελειώνει η θητεία του Κοινοβουλίου και θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε προσωπικά ως Πρόεδρο που μας φέρατε σε αυτό το <laughs> τέλος της θητείας, ε, σοους και αυλαβής και πάντα με μεγάλο κύρος, καμιά φορά και με πίεση. <laughs> Ξέρω, πιεζόμαστε πολύ και εμείς καμιά φορά, εσείς ακόμα περισσότερο και στην πατρίδα σας ίσως είχατε κάποιες προσωπικές ε, δυσκολίες. Αυτό μπορεί να συμβεί στον οποιοδήποτε. Πάντως σας ευχαριστώ προσωπικά και Δημόν, τη Γραμματεία και τον Αντιπρόεδρό σας ή τους Αντιπρόεδρους σας που αναλάβαναν την Προεδρία όπου τελείπατε. Λοιπόν, και εμένα η τελευταία φορά που μιλάω στο Κοινοβούλιο, εκτός αν έχετε άλλα σχέδια ε, μυστικές συναντήσεις και τέτοια. Τελευταία επίσημη ε, συνεδρίαση μετά από 10 χρόνια αποχωρώ κι εγώ. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους, ήταν πολύ καλοί συνάδελφοι. Και ήταν ε, επικοδομητική η Επιτροπή πάντα και ευχάριστη. Να σκεφτούμε τι περάσαμε τώρα τις κλιματικές αλλαγές και κάποια άλλα θέματα, διασυνοριακή περίθαλψη. Είναι μεγάλα θέματα και καταφέραμε ως Επιτροπή να το κάνουμε. Σας ευχαριστώ όλους, μέλη, βοηθούς, το προσωπικό, τους διερμηνείς στην επιμελητία. Όλοι αυτοί που φροντίζουν να έρχονται εδώ κομμένα δέντρα στα γραφεία μας και μετά να μαζεύουν τα χαρτιά που αφήνουμε. Τα λέω έτσι με μεγάλη ζέστη, ζέση και εύχομαι κάθε επιτυχία στους συναδέλφους και να έχετε υγεία, ευτυχία και χαρά στο Νέο Κοινοβούλιο. Σας ευχαριστώ. Yeah, thank you very much. Σας ευχαριστώ πολύ, Τζον. Ό,τι καλύτερο και για σένα, από όλους μας. Ο Γκουίντο Θα κάνω mm, ακριβώς αυτό που έκανε ο Τζον Bowes πριν. Συμφωνώ. Συμφωνώ. Σόνο Συμφωνώ ε, για τα όσα είπε για τον ε, αμίαντο, λέω και εγώ τα ίδια. Λοιπόν, θα μπορούσαμε ίσως να τελειώσουμε με δάκρυα στα μάτια. Ε, είμαστε σχεδόν έτοιμοι να ξεγλιστρήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Λοιπόν, και για μένα ήταν εξαιρετική αυτή η εμπειρία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους σας, όλους τους πρωταγωνιστές και εσάς ιδιαίτερα κύριε Πρόεδρε. Ε, πραγματικά δεν ήταν εύκολες, ε, εύκολα τα πρώτα βήματα αυτής της Επιτροπής. Ε, δεν ήταν εύκολο αυτό το πέρασμα, είχαμε να αντιμετωπίσουμε δύσκολα εγχειρήματα, εσείς τα καταφέρατε, κρατήσατε πραγματικά τις ισορροπίες, ε, το κάνατε με πολύ σωστό τρόπο και βεβαίως είχατε να αντιμετωπίσετε μεγάλες δυσκολίες το παγκόσμιο ρεκόρ ταχύτητας στην λήψη αποφάσεων σχετικά με προτάσεις νομοθετικού περιεχομένου και βεβαίως οι διπλωματικές σας ικανότητες και λοιπές σας ικανότητες ε, εκτιμήθηκαν ιδιαίτερα. Ε, θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω και όλους τους συναδέλφους και βεβαίως δεν πρέπει να παραλείψω τη γραμματεία η οποία έπαιξε έναν αποφασιστικό ρόλο. Ε, ε, και μετά θα πάμε να πιούμε ένα ποτηράκι έτσι. Νομίζω ότι δεν μπορούμε να τελειώσουμε έτσι. Ε, πρέπει να υπάρξουν και αποχαιρετισμοί και νομίζω ότι θα πρέπει επίσης να αναγνωρίσουμε τη συμβολή των διερμηνέων γιατί κάνουν πολύ σημαντική δουλειά. Και βεβαίως η συμβολή τους είναι αποφασιστική σημασίας. Λοιπόν, Λοιπόν, το, τα αγγλικά του Ρίτς τα ξέρω απ' έξω, απ' έξω και με τέλεια, τέλεια. Ε, αλλά για να πω μπονασέρα, καλησπέρα, έχω μερικές δυσκολίες στα αγγλικά. Thank you very much indeed. Chris Davis. Ευχαριστώ, Chris Davis. Πολύ σύντομα, Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ενώσω τη φωνή μου με τις ευχές και τις ευχαριστίες προς το προσωπικό του Διερμηνής και σας προσωπικά. Ξέρω ότι έχετε και το θάρρος της γνώμης σας και είχαμε την ευκαιρία να σας ακούσουμε επανειλημμένα. Τα τελευταία δυόμιση χρόνια χάρηκα που δεν συμφωνήσατε ποτέ με την Κάρολάιν Τζάξον που συστηματικά υποτιμάει τους φιλελευθέρους. Ε, Πράγματι είχατε πνεύμα δικαιοσύνης και επικοδομητικό και πάντα θέλετε να εκπροσωπείτε ως πρόεδρος της Επιτροπής μας στην Επιτροπή στο Κοινοβούλιο εξάρτητα από την πολιτική σας ομάδα και τις πεπιθήσεις σας. Ευχαριστώ. Thank you. Thank you very much. Very much Ευχαριστώ πολύ. Ο Σλούτερ. Yeah, I must say also that you us in the... Θα ήθελα να σας πω ότι και εμείς ανησυχούσαμε λόγω αυτού, οι πράσινοι, ε, αλλά δεν ε, συνειδητοποιήσαμε ότι τελικά δεν είχαμε δίκιο και εκτιμούμε την προεδρία σας. Μπόβις, ε, έκανε ένα πάρα πολύ ωραίο λόγο και απλά θα συμφωνήσω μαζί σου. Ένα. Ο Μπλόκλαντ και μετά η Ντάκμαρ Μπέρετς. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και για μένα η τελευταία συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος. Μετά από 15 χρόνια δούλεψα με πολύ μεγάλη ευχαρίστηση και κέφι και όπως και ο Γκουίντο και ο Τζον θα εγκαταλείψω την Επιτροπή αυτή. Πρέπει να σας πω ότι τα τελευταία πέντε χρόνια ήταν τα πιο ενδιαφέροντα της 15 ετίας. Κάναμε τρομερή δουλειά. Πάρα πολύ νομοθεσία πέρασε την τελευταία πενταετία και ε, πιστεύω ότι σε ό,τι μας αφορά η Επιτροπή Περιβάλλοντος δούλεψε πάρα πολύ καλά και πρέπει να σας πω ότι τα τελευταία μισή χρόνια από τη δική σας Προεδρία είχα καμιά φορά ε, περισσότερο την ευκαιρία να κάνω μερικά πράγματα από ό,τι στο προηγούμενο διάστημα om eh, samen met u... Και πραγματικά το βρήκα πολύ ευχάριστο αυτό. Είχα την ευκαιρία να εκπροσωπώ την Επιτροπή Περιβάλλοντος όταν εσείς ήσασταν σε κανένα αεροπλάνο ή δεν είχε απογειωθεί καθόλου και τέτοια και να λάμβανα εγώ τα καθήκοντά σας. Το θεώρησα πολύ ευχάριστο λοιπόν και συνεργασία με τη Γραμματεία και τους ε, διερμηνείς που πάντα μας βοηθούν, τους συνεργάτες ε, των συναδέλφων πάντα είχαμε άριστη συνεργασία με όλους. Αυτό νομίζω είναι πραγματικά χαρακτηριστικό της Επιτροπής Περιβάλλοντος. Προσπαθούμε να κάνουμε καλύτερο το περιβάλλον, το κλίμα και πιο υγιεινό. Νομίζω ότι ήταν κοινή μας αφετηρία και πάντα ήταν πολύ ενδιαφέρον για μένα. Ελπίζω να μην ε, χαθούμε, δεν θα μολύσετε πάρα πολύ. Μένω και κοντά, Σε λίγα χιλιόμετρα μας χωρίζουν, θα τα ξαναπούμε. Thank you very much, Hans Ευχαριστώ πολύ, Hans. Η κυρία Ντάγμα Ροτ Μπέρεντ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Στα αγγλικά. Συνήθως είμαι πάρα πολύ προσεκτική με την ετικέτα και το πρωτόκολλο. Δεν μπορώ να μιλάω μετά τον ε, συντονιστή μου, αλλά ας κάνω μια εξαίρεση σήμερα για αλλαγή. Εγώ αισθάνομαι εδώ πολύθωμα κοιτάζοντα γύρω γύρω. Είμαι 20 χρόνια στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και από τα 20 χρόνια 15 ήμουν συντονίστρια στην Επιτροπή του εδώ. Την τελευταία πενταετία ανέλαβε ο Γκίντο. Με θαυμάσιο τρόπο. Εγώ θα ξανάρθω ε, στο επόμενο κοινοβούλιο. Ξέρω ότι είναι δύσκολο για μερικού να το πούνε, αλλά με το γερμανικό σύστημα το ξέρω ότι θα ξανάρθω. Δεν είναι γεγονό. Κανένα δεν χαίρεται όταν τον αλλάζουν. Ήταν αρχικά πρόεδρος ο Καρλ Χάιντ Φλόρενς, ε, τον γνωρίζαμε, δεν θέλαμε να χάσει τη θέση του και ο Γκίντο και εγώ, αλλά πραγματικά πρέπει να πω ότι ε, σας αναγνωρίζω ότι εσείς κάνετε πολύ καλή δουλειά, πολύ δίκαιο πάντα, ε, με μεγάλη διαφάνεια και ε, συμπεριλαμβάνατε τους πάντες. Και πραγματικά μου άρεσε πάρα πολύ ο τρόπος με τον οποίο προεδρεύατε. Δεν έχω τίποτα να ε, σε επικρίνω παρά να σας πενέσω. Ομάδα ήταν ε, και ο κ. Χούμπε και κάποιοι άλλοι άλλαζαν. Γιατί πήρα το λόγο λοιπόν. Βεβαίω θέλω να ευχαριστήσω του Διερμηνεί που ελπίζω να του δούμε όλου ξανά μετά τον Ιούλιο. Αλλά δεν γνωρίζουμε πολλά πράγματα, δεν γνωριζόμαστε καλά μεταξύ μα. Εγώ δεν ξέρω αν κατεβαίνει κανεί ξανά, τι κάνει στη ζωή του, τι σχέδια έχει, με το πάω μέχρι εκεί. Για κάποιου συναδέλφους δεν ήξερα καν αν θα είναι πάλι υποψήφιοι, αν θέλουν να επανέλθουν για τον Κρίντο, το ήξερα. Μου είχε πει νωρίτερα ότι έχω και άλλη ζωή εκτός από εδώ μέσα. Έχω και άλλα πράγματα στη ζωή μου εκτός από το κοινοβούλιο. Εγώ <laughs> τον βλέπω να ε, πεζοπορεί εκεί κάπου στη Φλωρεντία και στους λόφους από πίσω στη Δοσκάνη. Μια χαρά ε, θα είναι ε, στην υπηρεσία στο Ελσίνκι για ε, τη χημία. Εγώ θα μπορούσα να προτείνω και άλλα. Όταν παίρνει τέτοιο ύφο, άσε καλύτερα. Θα τα πούμε άλλη στιγμή αυτά. Και ήξερα από τον Τζον Μπόις τι είπε και αυτός ότι έχω και άλλη ζωή και όλοι μας άλλωστε. Μπορεί να ξέρετε τη φράση αυτή που λέει ότι η ζωή ε, ε, ένα έτος στη ζωή του σκύλου αντιστοιχεί σε 7 χρόνια ανθρώπινη ζωής. Ε, το βουλευτή αυτό διπλασιάζεται. Μέχρι χθε δεν ήξερα ότι δεν θα ξανάρθει το ΡΕΤ. Για τους άλλους, δηλαδή, ο κύριος Αδάμου ας πούμε και κάποιοι άλλοι, δεν ήξερα καν ότι ο Χάνς Μπλόκλαντ φεύγει τώρα μόλις το, αυτό το δευτερόλεπτο. Καμιά φορά δεν έχουμε ούτε το καιρό να συζητήσουμε. Θα είναι αλλιώ τα πράγματα και η δουλειά πολύ διαφορετική. Πραγματικά εκτιμώ όλη τη δουλειά που κάνατε εδώ. Δεν ήταν πάντα εύκολη. Δεν είχαμε πάντα τι ίδιε απόψει, ούτε καν η Ντορέτ και εγώ α πούμε. Αλλά είχαμε την αμοιβαία κατανόηση ότι θέλαμε να φτάσουμε σε συμβιβασμό. Έστω και στο εσωτερικό τη δική μα ομάδα και καμιά φορά και με άλλε ομάδε. Και αυτό έκανε τη δουλειά μα τέτοια ευχαρίστηση και τόσο κέφι. Θα μου λείψετε πάρα πολύ. Θα καθυστερήσω. Γιατί είχα κανονίσει κάτι άλλο, έμαθα ότι στις 6.30 κερνάτε. Εντάξει, θα έρθω εδώ. Δεν θέλω να βουρκώσω και να κλάψω, αλλά όσοι ξανάρθετε και ε, θα έχουμε επιρροή. Αλλά όλοι γνωρίζετε πώς δουλεύει η Επιτροπή αυτή και τι μορφή έχει και πώς συμπεριλαμβάνει τόσα πολλά θέματα, πόσο δύσκολο μπορούν να διαχωριστούν τα θέματα. Αυτά είναι αλληλένδετα, σαν πάζελ συνενώνονται, σαν ψηφιδωτό. Παρακαλώ θυμηθείτε το αυτό, θα ζητήσει η πολιτική ομάδα σας, ε, διάρθρωση επιτροπών και τα λοιπά συμπαρμαρτούντα, γιατί πολύ συχνά ακούμε πολλές επιθυμίες και πολλές επιβουλές. Και η επιτροπή μας δεν ήταν πάντα η πιο αρεστή με τον τρόπο που δούλευε σε όλες τις πολιτικές ομάδες. Ακούμε διάφορες φήμες ήδη στους διαδρόμους. Και οι φήμες αυτές δεν είναι από φίλους του Κοινοβουλίου, ούτε απαραίτητα φίλους της Επιτροπής μας. Παρακαλώ θυμηθείτε και μην το ξεχνάτε αυτό το πνεύμα στο οποίο συνεργαστήκαμε και όλοι αυτοί που δεν θα επανέλθετε. Ελπίζω να δείτε ότι υπάρχει και άλλη ζωή εκτός Κοινοβουλίου που είναι τόσο ευχάριστη. Ευχαριστώ. Thank you very much indeed to all of you and uh, to all the members. Σας ευχαριστώ και ευχαριστώ όλα τα μέλη της Επιτροπής θα ήθελα να σας πω κι εγώ κάποια λόγια. Για μένα ήταν πολύ θετική η εμπειρία. Σας ευχαριστώ όλους για τη συνεργασία σας. Σας ευχαριστώ για όλες τις μέρες όπου δίπλα σας έμαθα πώς είναι να προεδρεύει κανείς σε μια επιτροπή, να δουλεύει στο κοινοβούλιο, Έχω μια πολιτική σταδιοδρομία, ένα χρόνο έμεινα παρατηρητής και αυτή η καλή εμπειρία ήτανε. Και όταν έγινα αντιπρόεδρος μαζί με την Ντάγμαρ, θεώρησα ότι είχα φτάσει στο απόγειο της ε, σταδιοδρομίας μου, αλλά τελικά ε, έγινα και πρόεδρος επιτροπής μετά. Αυτό είναι το απόγειο της καριέρας μου είναι αυτή η θέση, αυτό το αξίωμα ε, με κάνει να νιώθω επιτυχημένος. Έζησα και κάποια προσωπικά δράματα βέβαια, δεν μην υπερβάλλω, δεν ήταν δράματα. Αλλά τέλος πάντων γενικά είναι καλή αυτή η πολιτική στα διαδρομιά. Θα προσπαθήσω να επιστρέψω. Ε, θα καταβάλω κάθε δυνατή προσπάθεια. Δεν νομίζω να ξαναγίνω πρόεδρος. Ε, γιατί δεν θα έχει την ίδια επιτυχία το κόμμα μου. Ξέρετε πώς είναι η μοιρασιά ανάμεσα στι πολιτικές ομάδες. Αλλά υπόσχομαι ότι αν τελικά επιστρέψω θα προσπαθήσω να είμαι στην Επιτροπή Περιβάλλοντος και να συνεχίσω τη δουλειά αυτή, να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε. Σας ευχαριστώ πραγματικά και ε, σας περιμένω το βράδυ, ελπίζω να σας δω. Α, και μην ξεχάσω, ευχαριστώ τον Άντρα Ζούμπερ και το λοιπό προσωπικό, ο Ανδρέας, ήταν ο φύλακας άγγελός μου, ήδη από την αρχή. Και δεν θα ήμουν τόσο καλός πρόεδρος όπως εσείς το θέσατε δηλαδή χωρίς αυτόν. Σας ευχαριστώ. Θα κλάψω. Δεν ήταν κακό. Τώρα, έχουμε κάτι συντονιστές σε λίγο για κάποια τεχνικά θέματα που πρέπει να αποφασίσουμε και νομίζω θα τελειώσει σύντομα για αυτή η συνεδρίαση.